El señor presidente. Καλή σα ημέρα, φίλε και φίλοι. Κυρίζω την έναρξη τη ε, Συνόδου για σήμερα Πέμπτη. Μετά από το χθεσινό αγώνα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται την έκθεση του κυρίου George Lyon σχετικά με το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ο Επίτροπος βρίσκεται ανάμεσά μας διότι γνωρίζω πως ε, αυτή την ε, εβδομάδα ε, Συναντήσαμε πολλούς επιτρόπους, αλλά δεν ήταν πάντα οι αρμόδιοι επί των θεμάτων που εξετάζαμε. Και στο στην περίπτωση αυτή έχουμε τον αρμόδιο επίτροπο και αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο πρωτίστως στον κύριο George Lyon, ο οποίος ως συγητής αυτής της σημαντικής έκθεσης θα μας μιλήσει για τέσσερα λεπτά προκειμένου να παρουσιάσει την έκθεσή του και δύο λεπτά για να απαντήσετε στο τέλος της συζήτησης. Ο εισηγητής φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα έξι λεπτά στην αρχή του παρουσίαση, αλλά τότε θα το επομένει χρόνος προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέλφων και στους σχολιασμούς σου. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να χρησιμοποιήσει τα τέσσερα λεπτά αρχικά. Εν είναι κυρίως του εαυτού του και θα κάνει όπως νομίζει. Κύριε Λάιον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ε, προσφέροντας τα συλληπιτήριά μου και τα συγχαρη... στους Γερμανούς συναδέλφους και τα συγχαρητήρια στους Ισπανούς συναδέλφους μετά από τον εξαιρετικό αγώνα. Θέλω να ξεκινήσω με τα δύο βασικά θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε από πλευράς της αναθεωρήσεως της ε,